κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 141, ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίφτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα αρχίζει η ψηφοφορία Πέρασα. 27-29 απερίφθη. Και τρεις αποχές. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Ξανά. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Θέλετε έλεγχο για την 154. Πάμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αφού εγκρίθηκε, γιατί θες έλεγχο. Λοιπόν, 154. Πέρασε 42 ναι. υπέρ 16 κατά. Σαφές ήταν. 155 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. 67 συγγνώμη. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφτεται. Η συμβαστική 20. Τσεκ, τσεκ. Ελάτε τώρα. Ε, όχι. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 187. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ Α, τέσσερα, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος, είπα 44, τέσσερα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πέντε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έξι υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχο ε, έλεγχος παρακαλώ. 22-38 απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και το σύνολο λοιπόν τώρα ηλεκτρονικά για το κείμενο που στροποποιήθηκε. Die Abstimmung. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 56 υπέρ 6 κατά με καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Christian, who uh, represents Mrs. McAvoy. Ο Κρίστιαν ε, Πρέντα εκπροσωπεί την κυρία Μακοβέη. Ποιος. Με μεγάλη χαρά. Πάμε στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τώρα. Η 34 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 95 τμήμα δεύτερον. Ψήφι πέ. Κατά. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Έτσι, απερίφθη. Τσεκ. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει. Die ε, 17 υπέρ 38 κατά απερίφθη. Η τροπολογία 96 τώρα του κυρίου Νάρντ υπέρ της 96. Υπέρ της τροπολογίας λέγω 96. Κατά. Εγκρίνεται.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 103 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 ειπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 τώρα είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για πάμε στην 156. υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα της 164 ψηφίζουμε. Το δεύτερο, προσοχή, είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. Και το τρίτο τώρα. Έχει και τρίτο. Α, καταπίπτει, καλά. Πάμε στην 167 το είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 7 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 173. Έτσι, 173 Είπε Κατά αποχές εγκρίνεται 178 Είπε Κατά αποχές έλεγχος. Με την 178. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί όμως. Πέρασε. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 26-26. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 213 υπέρ κατά εγκρίνεται τσεκ 213 μα νομίζω ότι της δικής σου ομάδας ήταν Είμαστε στην τροπολογία 213. Πέρας. Εγκρίνεται 27 υπέρ 26 κατά. ...215, 16 και 18 υπέρ. Α, όχι, ξεχάσαμε τη 214, δεν καταπίπτει. Όχι, όχι, 13 εγκρίθηκε, όχι 12. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη 214 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκε. Μόνο το ΕΛΚ καταψήφισε. Ναι. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. 214 αρχίζει η ηλεκτρονική απολύθευση. Πέρασε. 23 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. Πώς είπατε. Και εμείς όλοι από εδώ κατά ψηφίζαμε, αλλά δεν κοιτάτε προς τα δω ωραια Ωραία, 23-29 απορρίπτεται. Τι πρόβλημα έχετε ακριβώς. I think I was 10 times right and one time wrong. Εντάξει, 10 φορές εδώ βρήκα και μια φορά έπεσα έξω. Ε, καλή αναλογία είναι 10 προς 1. Δεν χρειάζεται να μου τα λέτε τόσο έντονα. Λοιπόν, 215, 216, 218. Μαζί. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 217 Ειπέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 211 war angenommen, nein. Wir kommen zu 219. 219 ειπε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 ειπε Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για να δούμε τι γίνεται με το 220. Άρχεται η ψηφοφορία. 20 υπέρ, 33 ε, κατά απορρίπτεται, 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ, 228 υπέρ, κατά, υπέρ πρώτα, κατά, αποχές, έλεγχος. 228. Πέρας. Απορρίπτεται 15 υπέρ 26 κατά. 230 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Απόχες. 232 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 233 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πού πάμε. 237 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 239 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 240 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 241 υπέρ, 51 συγγνώμη, κατά, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 251. Πέρας. 24 υπέρ, 25 κατά και 5 εποχές. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 265 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 266, 267, 268 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 269, έτσι δεν είναι, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 273 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 275 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 277 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 278 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 είπε όχι. 279 πρώτα είπε κατά αποχές. Εγκρίθηκε η τροπολογία του παρόλο που ο ίδιος ο κύριος Χάουιτ δεν ψήφισε. Συμβαστική 15 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 280 είπε. Κατά. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί, αλλά να το δούμε. 280. Πέρασε. Εγκρίθηκε 24-22. 282 υπέρ κατά άποχες απορρίψετε. Συμβαστική 16 16π. Κατά άποχες εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε. Πώς είπατε, Κρίστιαν και εσύ θες τώρα στοίχημα ένα διπλό ουίσκι. Ωραία, πάμε. Ας το ελέγξουμε. 292 ηλεκτρονική υπορρίθευση. Τζέιμσον με πάγο ή χωρίς πάγο. Καλά, θα δείξει. Πέρασα. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Ω. Oh. Χωρίς πάγο τότε. 293 dafür. 293 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26, 27, 28, 29, 30. Κάποιος έχει πολλούς φίλους εδώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά όχι αρκετούς μάλλον. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 μέχρι και 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψει. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψεται. 50 μέχρι και 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-46 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64-44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία τώρα 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Ναι, Κριστιαν. Να ψηφίζει η ομάδα σου. Τι να σου κάνω. Άρχεται η ψηφοφορία. Που είμαστε στην 65. Λοιπόν, πέρας, είναι τη σχέση Μακοβέη. 18 υπέρ 36 κατά απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 όχι έχει διεκπεριωθεί και πάμε στην 69 όχι στην 70 70 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 έως 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 μέχρι και 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, πρέπει να ψηφιστεί και 72. Ναι, εγώ σας το έλεγα όμως. Ε, ξεχάσαμε την τροπολογία 72 γιατί οι προηγούμενες απερίφθησαν. Πρέπει να ψηφιστεί υπέρ της 72. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οι δύο τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία βαρθών 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21-27. Και καταπίπτουν οι δύο επόμενες και πάμε στην 5 μέχρι και 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 με 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 17 με 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 είναι γλωσσική υπόθεση. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία η οποία αρχίζει αυτή τη στιγμή. Die Abstimmung ist Εγκρίθηκε η έκθεση με 47 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Πρέντα. Κύριε Μάκουβάη δηλαδή. Βάιγγελ. Βάιγγελ είναι λέει ο Πρέντα. Εντάξει, Βάιγγελ. λοιπόν, επόμενη, η Σερβία. David Μακάλιστερ εισηγητής. Έχετε να δηλώσετε τίποτα? Όχι. Πάμε λοιπόν. Τροπολόγια 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η προφορική 3. Κύριε Χάουιτ, ναι, συγγνώμη. Όταν ε, ανοίξαμε τη συζήτηση από χτε, ε, συζητήσαμε με τι ομάδε πριν την Ολομέλεια. Δεν υποστηρίζουμε όμω ε, αυτή την τροπολογία. Ωραία, συμβαστική 4. Διαφωνείτε με την προφορική. Πάμε στην επόμενη. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ 41. 41, εντάξει, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η συμβαστική 6 υπέρ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 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. Η συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 131, τμήμα πρώτον. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 30-26. Συμβαστική 15 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 146 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166-167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ωραίο ζευγάρι 68. 158 λέει ο πρόεδρος. Κατά, εγκρίνεται. 159, συγγνώμη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 160. Θα πρέπει λέει να ψηφιστεί με την προφορική τροπολογία παριθμών 1, η οποία που είναι όμως. Ψηφίζεται υπέρ αυτής της τροπολογία μαζί με την προφορική 1. Εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 175 σε τμήματα. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 21 κατά και αποχές εγκρίνεται. 186. Τμήμα πρώτον. Ψήφι π. Κατά αποχές εγκρίνεται. 187 Επέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 188 Επέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 188. Επέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205 η τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερθών 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 και 10 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 14 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 12 και 15 μαζί είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 έχει καταπέσει. Λοιπόν, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο αρχίζει τώρα. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Δεν ήταν και τόσο τραγική η ε, διαφορά. 50 υπέρ, 4 ε, κατά και 2 εποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Λοιπόν, θα διακόψουμε τώρα τη συνεδρίαση για 25 λεπτά. Λίγο πριν τις 11 να ξαναρχίσουμε για την ακρόαση. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι μπορειογνώμονες. Ελπίζω να παραμείνουν οι συνάδελφοι βέβαια στις 11. Λοιπόν, καλό καφέ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 Υπότιτλοι capable de Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε θερμότατα στην ακρόασή μας. Η αφορμή ε, είναι η προετοιμασία της, ε, και εκπόνηση της έκθεσης του συναδέλφου Γκαμπριέλου Λαντσμπέργης για τη σχέση μας με τη Ρωσία. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η σημασία αυτού του θέματος, διότι οι σχέση μας με τη Ρωσία ενδεχομένως να βρίσκονται σε καμπή, αν κοιτάξουμε και τις εξέλιξεις στην Ουκρανία. Για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ναι καθεν ήταν ξεκάθαρο ότι πρώτον θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία και δεύτερον οι σχέσεις αυτές για τη Ρωσία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ήταν πάρα πολύ θετικές εάν ο καθένας στηρούσε τους κανόνες. Διαπιστώνουμε ότι με την προσάρτηση της Κρυμαίας και με τη ρωσική συμμετοχή και τη στρατιωτική και με προσωπικό και με όπλα στην Ανατολική Ουκρανία παραβιάζεται ε, το διεθνές δίκαιο. Και η εδαφική ακαιρεότητα της ε, χώρας και η αυτοδιάθεση των λαών και η κυριαρχία δεν γίνεται σεβαστή. Με περίεργο τρόπο λοιπόν εκεί ορίζουν το διεθνές δίκαιο. Στο Μόναχο είχα μια μικρή αντιπαράθεση με τον κύριο Λαυρόφ όταν άκουσα πώς ορίζει εκείνο το διεθνές δίκαιο, ότι επιτρέπεται δηλαδή να παραβιάσεις τα σύνορα μιας άλλης χώρας όταν θεωρείς ότι έχεις ιστορικές αξιώσεις και υποτίθεται ότι θέλεις να προστατεύσεις εκεί μειονότητες. Αυτό είναι ορισμός διεθνούς δικαίου. Με θερμινευόμενο αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρα ε, έχει ε, θεμητό δικαίωμα να ε, επεμβαίνει σε μια άλλη. Εγώ έχω γνωρίσει εποχές στην Ευρώπη και τέτοιες που έχουν να κάνουν σχέση και με τη δική μου χώρα που χρησιμοποίησαν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Και εμείς θεωρούσαμε ότι αυτά τα επιχειρήματα στην Ευρώπη πλέον έχουν εκλείψει ότι με την τελική πράξη του Ελσίνκη και το χάρτη των Παρισίων και όλα τα συμπαρομαρτούντα που ακολούθησαν και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση το μνημόνιο της Βουδαπέστης δεν υπάρχει πλέον λόγος να παραβιάζεται η εδαφική ακεραιότητα και η ε, κυρίαρχη απόφαση κάθε λαού για το τι συμβάσεις και συνθήκες θα υπογράψει. Και επαναλαμβάνω, αν δεχόμασταν τα τρία αυτά σημεία, Μπορεί ο καθένας που έχει ιστορικούς λόγους να μπαίνει σε μια χώρα να μπαίνει όταν λέει ε, παραβιάζονται ή απειλούνται δικαιώματα μειονοτήτων. Ή είναι τόσο τεράστια η ευαισθησία του καθενός ε, και τα άχη και αγωνίες που θέλει να τα ε, κατευνάσει. Αν πηγαίναμε έτσι θα μπορούσα να σας αναφέρω και 100 σημεία στην Ευρώπη όπου θα ξεσπούσε πόλεμος. Αυτά τα θέματα μας απασχολούν πολύ. Πρέπει να σας πω επίσης ότι με μερικά μέλη της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο πήγαμε και είχαμε ένα πρόγευμα με το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το ρωτήσαμε αν υπάρχει έστω και μία περίπτωση ε, στο ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης ή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου οι ρωσόφωνοι, οι ε, ρωσο, ρωσογενείς της Ουκρανίας ή ε, η ίδια η Ρωσία να έχει προσφύγει λόγω διακρίσεων κατά των ρωσοφόνων ή ρωσογενών ε, στην Ουκρανία. Και μας είπε ότι δεν υπάρχει παραμικρή υπόθεση ούτε στο δικαστήριο ούτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μηδέν. Δηλαδή αυτά που λέει η προπαγάνδα Βεβαίω έχει δικαίωμα, η Ρωσία είναι μέλο του Συμβουλίου τη Ευρώπη και μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και στην υπουργική διάσκεψη. Έχει μάλιστα και δικαστές αποσπάσει. Υπάρχει ο ΣΑ, υπάρχει το Συμβολίο της Ευρώπης και μια σειρά θεσμών που έχουν δημιουργηθεί για να λύνονται αυτά τα προβλήματα ειρηνικά και δεχόμενε συγκρούσεις να προλαμβάνονται και να μην ε, παραβιάζει κανείς την εδαφική ακεραιότητα κανενός μονομερός. Και δεν τα χρησιμοποίησε η Ρωσία που είναι μέλος και στον ΟΑΣΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και ε, είναι και εύλογο αυτό γιατί δεν στέκουν οι ισχυρισμοί τη, δεν θα έστακαν στο δικαστήριο. Και επανέρχομαι λοιπόν στην πρώτη πρόταση ότι καλό θα ήταν και λογικό και οι δύο πλευρέ να έχουν σχέση καλή γειτονίας. Και οικονομικά και πολιτικά είναι αυτά σημαντικά και τις επόμενες μέρες θα δούμε τι θα βγει από τη Συμφωνία Μίνσκ 2. Υπάρχουν και καλές και κακές ειδήσει. Υπάρχουν και η τρίτη κατηγορία, οι χείριστες ειδήσει. Ε, δεν ξέρουμε μέχρι πού θα κλιμακωθεί αυτό, γιατί ορισμένα έχουν παραβιαστεί, ιδιαίτερα σε ένα σιδηροδρομικό κόμβο. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα πρέπει όμως το εξή να είναι πάρα πολύ σαφές, ότι για να λειτουργήσουν όλα αυτά η Ρωσία θα πρέπει να αναγνωρίσει δημοσίως ότι είναι τμήμα της σύραξης, εμπόλεμο ε, ε, ε, παράγων. Αυτό εν μέρη το αναγνώρισε στο Μίνσκ, αλλά για να λυθεί το πρόβλημα θα πρέπει η Ρωσία να, αναγνωρίσει και δημόσια ότι συμμετέχει στη μάχη και όχι απλώς συνοδεύει ή πελεσιώνει μια άλλη εμπόλεμη πλευρά. Για μας αυτά είναι πολύ σημαντικά. Χαίρομαι που και μετά από ε, τη δράση του κυρίου Λαντσμπέργης έχουμε τρεις ε, εγνωσμένου κύρους ε, γνώστες πραγματικά της κατάστασης και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να Καλωσορίζω την κυρία Μαρή Μεντράς από το Πανεπιστήμιο τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παρισίου, ε, τον κύριο Μόσες ε, από ε, το Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων του Ελσίγη και τον κύριο Φόρμπιχ από το γερμανικό Marshall Fund του Βερολίνου. Και με αυτή τη σειρά θα σας πρότεινα να ξεκινήσουμε και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μαρή Μεντράς. Σας παρακαλώ. Α, ξέχασα τον κύριο Λαντσπέργης. Ναι, ίσως να κάνει και αυτός μια σύντομη εισαγωγή. Θα κάνει και ε, σύνοψη στη συνέχεια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ομιλητές που βρήκαν το χρόνο στο πολύ βεβαρημένο τους χρονοδιάγραμμα να έρθουν για να μας, να μας μιλήσουν και να εκφράσουν την άποψή τους για ένα από τα πιο σημαντικά πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα της εποχής μας, οι ευρωρωσικές σχέσεις. Όταν ξεκίνησα τη σύνταξη αυτής της έκθεσης, πολλοί με τους οποίους συναντήθηκαν μου είπαν ότι επρόκειτο για κάπως αδύνατη αποστολή το εγχείρημα να ορίσω τις ευρωρωσικές σχέσεις σε μια τέτοια εποχή, εποχή με τόσο μεγάλες αλλαγές και εξελίξεις. 44 χρόνια προσπαθούμε να καθορίσουμε τις σχέσεις ε Ρωσίας και δεν το καταφέραμε. Πώς θα το καταφέρετε τώρα. Στα τέλη του 2014 υπήρξε μια σχετική ηρεμία στην Ουκρανία και ε, θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να ανοίξει μια νέα, ε, να γυρίσει σελίδα η σχέση ε, ΕΕ Ρωσίας και θα πρέπει να ξαναεμπλακούμε με τη ρωσική πλευρά. Όμως με την έλευση του 2015 το τοπίο άλλαξε άρδιν. Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να καθορίσει τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ με τη Ρωσία. Και πράγματι είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό. Οι συμφωνίε του Μίνσκ 1 και 2 είναι ένα καλό παράδειγμα του πώ προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ρωσία. Είναι ο ευρωπαϊκό τρόπο να υιοθετήσουμε την προσέγγιση που θα βασίζεται στο κράτο δικαίου, να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να αρχίσουμε να συζητούμε, να μιλούμε για πράγματα. Όμω είναι δύο κόσμοι ξεχωριστοί αυτοί ο ένας κόσμος έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ελευθερία της έκφρασης και ο άλλος κόσμος έχει ένα τελείως διαφορετικό σετ εργαλείων που μπορεί να αξιοποιήσει και να χρησιμοποιήσει σε όποια κατάσταση φρονεί ότι είναι σκόπιμο να κάνει κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές υποθέσεις σε αυτό το κοινοβούλιο ήταν η υπόθεση της Ουκρανής πιλότου Σαφτσένκο. Η Ρωσία συνέλαβε ε, μία γυναίκα από το ουκρανικό έδαφος, την έβαλε φυλακή σε ρωσικό έδαφος, την βασάνισε και παραμένει εκεί τώρα. Και δεν θα αναφερθώ καν στις περιπτώσεις, στις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον ΠΟΕ και με την ε, υφαρπαγή γης στην Ουκρανία. Θεωρούμε ότι η Ευρώπη έχει μεταμορφωτική δύναμη. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να εμπλέξουμε τη Ρωσία ε, ότι μπορούμε να έχουμε συμβάσεις μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ λαών, μεταξύ επιχειρήσεων και ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα μεταμορφώσουν τη Ρωσία. Τίθεται το ερώτημα όμως, τα καταφέραμε, μπορέσαμε να το κάνουμε ή λειτουργήσε αυτό αντίστροφα. Ε, ξέρετε τρόπο να πιστεύω εγώ ότι η Ρωσία μας μεταμόρφωσε σιγά σιγά τα τελευταία νέα και οι τελευταίες εξελίξεις για ε, τις διάφορες χρηματοδοτήσεις ε, διαφορών κομμάτων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, υποθέσεις κατά τα καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποθέσεις περιορισμού ελευθερίας της, έκθεσης, της έκφρασης και ούτω καθεξής. αυτά είναι αυτά τα οποία μας μεταμορφώνουν σιγά σιγά. Πριν από λίγους μήνες ήμουν σε μια συνάντηση και μου είπε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος ότι πρέπει η Ρωσία να καταφέρουμε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανεξαρτήτως κόστους. Και νομίζω ότι αυτό καθόρισε τις ευρωρωσικές σχέσεις, αυτή η επιθυμία για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον ρώτησα όμως ποιος είναι αυτός ο οποίος θα στρώσει το τραπέζι. Γιατί ξέρετε, η εικόνα που έχω εγώ στο μυαλό μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται στο τραπέζι και περιμένει τη Ρωσία να έρθει να καθίσει δίπλα της. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Θέλουμε να βρούμε διπλωματικές λύσεις, θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τους διαφόρους κανόνες που έχουμε στη διάθεσή μας, όμως ε, η Ρωσία πρέπει τώρα να στρώσει το τραπέζι και εμείς να αποφασίσουμε αν θα θέλουμε και θα θελήσουμε να καθίσουμε δίπλα της σε αυτό το τραπέζι εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Επομένως είναι πολύ σωστή η στιγμή να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση για τις ευρωβορωσικές σχέσεις. Δεν είναι μια αδύνατη αποστολή, είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να καθορίσουμε ε, τις ε, μελλοντικές εξελίξεις στο μέλλον των ευρωρωσικών σχέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Μέντρας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι μπορώ να είμαι εδώ και να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου για την κατάσταση έτσι όπως έχει σήμερα. Ο καθένας από μας έχει μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή του, 10 λεπτά εάν δεν τα πατώμε Και άρα πρέπει να διαλέξω τα σημεία στα οποία θα αναφερθώ και τα επιχειρήματα τα οποία θα προβάλλω. Σχολιάζοντας ε, την κατάσταση των ευρωρωσικών σχέσεων, των σχέσεων ΕΕ Ρωσίας. Πιστεύω ότι και οι τρεις μας θεωρούμε ότι το καθεστώς στη Ρωσία φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης για την υποβάθμιση των σχέσεων ΕΕ Ρωσίας, κυρίως λόγω της άμεσης επίθεσης, αν θέλετε, στα ανατολικά της Ουκρανίας και φρονούμε ότι οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας δεν μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα ακόμα και αν βρεθεί μια κάποια μορφή λύσης για το Ουκρανικό. Και το λέω αυτό διότι έχουν συμβεί πάρα πολλά ε, όπως το σχολίασε και μας το υποθύμησε και ο πρόεδρος Έλμαρ Μπροκ και ο ευρωβουλευτής ε, κύριος Λαντσπέργκης. Η ηγεσία της Ρωσίας έχει σύρει όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την ΕΕ ως φορέα, ως οργανισμό τους έχει όλους σύρει σε μια ε, κρίση ασφαλείας μεγίστου μεγέθους και χρειαστήκαμε αρκετό χρόνο για να το κατανοήσουμε αυτό, να το αντιληφθούμε ότι η ρωσική ηγεσία μεταμόρφωσε μια πολιτική κρίση ε, στην Ουκρανία ε, σε κρίση ασφαλείας τελικά ε, κατέρευσε το καθεστώς Γιανουκόβιτς Αυτή την, αυτό είναι ένα πολιτικό συμβάν η πτώση της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς και η Ρωσία το μεταμόρφωσε αυτό σε ένα μέγιστο ζήτημα ασφαλείας το οποίο εμπλέκει και αφορά τις περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρώπης και τον Ουκρανικό πληθυσμό βεβαίως. Το επιχείρημά μου λοιπόν είναι ότι η ηγεσία υπό τον πρόεδρο Πούτιν έκανε την επιλογή, διάλεξε να αντιπαρατεθεί με την Ευρώπη στο μέτωπο της ασφάλειας. Ε, η ρωσική ηγεσία προτιμά να υπάρξει αντιπαράθεση ε, ε, κυρίως και όχι τόσο διαπραγματεύσεις. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς, τους Ευρωπαίους, διότι θεωρούμε ότι οι δημοκρατίες έχουν, είναι καλύτερα εξοπλισμένες στο να διαπραγματεύονται, στο να βρίσκουν συμβιβαστικές λύσεις και θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ανταποκρίνονται στην ένοπλη παρέμβαση και στις αντιπαραθέσεις τέτοιου είδους, ειδικότερα όσον αφορά στην Ουκρανία η οποία δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία για 25 χρόνια έχει παραμείνει αν θέλετε κολλημένη, ε, τελματωμένη ανάμεσα σε εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ από τη μία και τη Ρωσία από την άλλη. Πρέπει να δούμε ποια απάντηση δώσαμε, πώς ανταποκριθήκαμε στη ρωσική αυτή πολιτική, ποια είναι τα διδάγματα που θα μπορούμε να αντλήσουμε. Από τις πρώτες απαντήσεις και αντιδράσεις που δώσαμε στην Ουκρανική κρίση θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό του πώς ανταποκριθήκαμε, να κάνουμε έναν απολογισμό τι μπορεί να κάνει ε, η Ρωσία και τι να μην κάνει ε, ε, σε επίπεδο κυβέρνησης και στρατού και ε, να κάνουμε έναν απολογισμό και μία αποτίμηση του κόστους όλων αυτών. Μπορεί κανείς να συγγράψει το αφήγημα της τελευταίας χρονιάς ως μία σειρά ρωσικών νικών. Έχουμε ρωσικές νίκες βάσει αυτού του αφηγήματος. Ένα άλλο αφήγημα όμως θέλει την τελευταία χρονιά να είναι μία σειρά ρωσικών λαθών αν υιοθετήσουμε άλλη οπτική γωνία και προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που δεν μπορεί να κάνει η ρωσική ηγεσία, δηλαδή να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, αυτό είναι το επιχείρημα που προβάλλω. Πολλοί συνάδελφοι έχουν διαφορετική άποψη για το πώς λειτουργεί η ρωσική ηγεσία και θεωρείται συχνά ότι ε, ο Πούτιν αρέσκεται περισσότερο σε κινήσεις τακτικής και δεν είναι τόσο μεγάλος στρατηγός. Εν πάση περιπτώσει, το δίδαμα που αντλούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτον ότι τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή, παρόλο που δεν είχαμε προβλέψει την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας από την Ρωσία και την περαιτέρω βία που ακολούθησε και παρόλο που δεν είχαμε προβλέψει και δεν περιμέναμε την πλατεία Μαϊντάν και την ειρηνική πτώση του καθεστώτος Γιανουκόβιτς και παρόλο που δεν είχαμε προβλέψει και δεν περιμέναμε την ικανότητα ε, των Ουκρανών να ακολουθήσουν το δημοκρατικό δρόμο με ελεύθερες και δίκαιες, νο, σύνομες αν θέλετε, εκλογές, παρόλα αυτά θέλω να τονίσω ότι οι Ουκρανικές αρχές δεν θέλησαν τη σύγκρουση, αναγκάστηκαν να ανταποκριθούν να απαντήσουν στην ένοπλη παρέμβαση και αποσταθεροποίηση του εσωτερικού της χώρους. Τα, παρόλα αυτά λοιπόν τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι ε, περιμέναμε λόγω του μεγέθους της κλίμακας της πρόκλησης αυτής και νομίζω ότι η ψήφιση των κυρώσεων εξέπληξε το Κρεμλίνο Άρα αυτό είναι ένα δίδαγμα που μπορούμε να αντλήσουμε στην προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια συνενετική και απλή πολιτική. Όταν έχουμε απλή συνενετική πολιτική, αυτή δουλεύει. Ότι δηλαδή η Ρωσία ε, έδρασε άσχημα, παράνομα και ως εκ τούτου μπορούμε να βρούμε ειρηνικούς τρόπους να εκφράσουμε την δυτική και ευρωπαϊκή άρνηση, απόρριψη τέτοιων ρωσικών μεθόδων. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και καλύτερα, ωστόσο. Εάν είχαμε καλύτερα πριν, ήδη πριν από αρκετά χρόνια καταλάβει και κατανοήσει τη φύση του καθεστώτος Πούτιν. Ότι δηλαδή είναι πολύ λίγες, ήταν πολύ λίγες οι επιλογές των Ουκρανών. με πολύ λίγες επιλογές θα κατάφερναν να πλοηγηθούν σε ειρηνικά νερά, συνεχίζοντας να ικανοποιούν να ευχαριστούν τη Ρωσία ενώ ταυτόχρονα ε, προσπαθούσαν να οικοδομήσουν ένα κράτος ε, δικαίου οδεύοντας προς την ευημερία και αποφεύγοντας ε, περαιτέρω πτώχευση και φτωχοποίηση. Ένα χρόνο μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις μας αμφιταλαντεύονται για άλλη μια φορά, υπάρχουν σημάδια κόπωσης του πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τον Πούτιν και αυτό κατά πάσα πιθανότητα εξηγεί τη Συμφωνία Μίνσκ 2 και πολύ φοβάμαι ότι όταν αμφιτελαντευόμαστε και δεν έχουμε σταθερά βήματα, επιστρέφουμε στην παλιά λογική μας, στην παλιά συλλογιστική, στους παλιούς φόβους και στην ανικανότητα του παρελθόντος. Για να αποφύγουμε λοιπόν κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να εξετάσουμε τη θέση της Ρωσίας, να την αντιληφθούμε όχι ως μία σειρά νικών από νίκες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τεράστιο τεράστιο κόστος της πολιτικής ε, που ακολουθούν στην Ουκρανία οι Ρώσοι. Έχει τεράστιο κόστος η, Ουκρανική, ε, η πολιτική του στην Ουκρανία για τη ρωσική οικονομία, κοινωνία ε, και ούτω καθεξής. Και τελικά θα τεθούν ε, τα ερωτήματα για, τις, για τους περιορισμούς στους οποίους θα προσκρούσει το ρωσικό καθεστώς όσο συνεχίζει με το πόλεμο στην Ουκρανία. Το κόστος της αντιπαράθεσης το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Το οικονομικό κόστος δεν είναι αμεληταίο. Δεν μιλούμε μόνο για τις κυρώσεις που έχουμε επιβάλει στη ρωσική πλευρά. Μιλούμε για αυτή την κληρονομιά ετών δυσλειτουργικής οικονομικής πολιτικής, οικονομίας που βασίζεται στους ε, και ε, ε, το κόστος της κατάρρευσης των τιμών πετρελαίου εδώ και τόσους μήνες. Ο Πούτιν ποτέ δεν μεταρρύθμισε πραγματικά τη ρωσική οικονομία. ανέκαθεν έδειξε την προτίμησή του σε ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα αυταρχικό και όχι απελευθερωμένο. Επομένως η κατάσταση στα οικονομικά είναι δεινή και η θέση της Ρωσίας είναι επιδεινωμένη σε όλους τους πολυμερείς οργανισμούς. Μεγάλο το κόστος που φέρει η ρωσική πλευρά λοιπόν. Το κόστος είναι μεγάλο και για το Κρεμλίνο, γιατί το, το Κρεμλίνο πόνταρε σε μια πιο εύκολη αποσταθεροποίηση ε, της Ουκρανίας και των νέων αρχών στο Κίεβο και τελικά ο Πούτιν έπρεπε να επενδύσει πολύ περισσότερο στο στρατιωτικό σκέλος από ό,τι είχε θελήσει και από ό,τι είχε προβλέψει. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα λοιπόν είναι αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι οι δυνατές επιλογές του Πούτιν, δεδομένου του ότι δεν έχει άπειρη άπειρους οικονομικούς, πολιτικούς ή στρατιωτικούς πόρους στη χώρα του. Εάν αξιολογήσουμε σωστά ποιες είναι οι δυνατές επιλογές, τι μπορεί τελικά να κάνει, ε, ποιες είναι οι ικανότητες της ρωσικής πλευράς σε πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό επίπεδο, τότε μπορούμε να διαμορφώσουμε καλύτερα τις απαντήσεις μας και άρα την επιρροή που μπορούμε να ασκήσουμε στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι Ρώσοι. Και τότε θα μπορέσουμε και καλύτερα να αποφασίσουμε ε, την διαμόρφωση των πολιτικών μας των δικών μας πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση γενικότερα ε, στην αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται η φύση του καθεστώτος στη Ρωσία. Δηλαδή αν η Ρωσία είχε μια κυβέρνηση πιο δημοκρατική που να σεβόταν περισσότερο το κράτος δικαίου, αυτή η Ρωσία θα ήταν σε θέση να δεχθεί την πλατεία Μάιντα, να δεχθεί την πτώση του καθεστώτος Γιαννουκόβιτς, να δεχθεί ε, κυβερνήσεις ουκρανικές πιο φιλοευρωπαϊκές και πιο ε, υπέρ μαχές αν θέλετε, οι υπερασπιστές της δημοκρατίας. Και ελπίζω να μην ξεχάσουμε το εξής ε, μάθημα πολύ γρήγορα. Αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί είναι ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι γέφυρα μεταξύ της Ρωσίας και ημών. Μια μεγάλη χώρα ε, σαν την Ουκρανία όπου ο πληθυσμός έκανε επιλογή την τελευταία χρονιά δεν μπορεί να κολλήσει να βρεθεί σε τέλμα μεταξύ μιας ρεβιζιονιστικής και αυταρχικής Ρωσίας από τη μία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη. Δεν είναι βιώσιμη λύση αυτό μακροπρόθεσμα. Τόσο απλά το λέω. Και δεν πρέπει να έχουμε τις ψευθεστήσεις σύμφωνα ε, με τις οποίες υποτίθεται η Ουκρανία μπορεί να είναι ουδέτερη. Γιατί αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θα είναι κυριαρχημένη από το μεγάλο της γείτονα. Και άλλωστε και οι άλλες χώρες της, που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς είναι μικρότερες, μεν, ωστόσο είναι άρεκτα συνδεδεμένες με το πολιτικό καθεστώς και τη δυνατότητα τους για οικονομική και άλλη ανάπτυξη. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οφείλουμε να προετοιμαστούμε για να αντιδράσουμε σε πολύ βραχυπρόθεσμες και άμεσες προκλήσεις και ανάγκες για λήψη αποφάσεων. Και αυτό να το συνδυάσουμε με μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική και τα δύο μαζί δηλαδή. Και να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε για για ό,τι μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη ρωσική ηγεσία και να στηρίζουμε την Ουκρανία όσο το περισσότερο μπορούμε, αλλά να προετοιμαστούμε ταυτόχρονα και για την Ρωσία μετά τον Πούτιν, γιατί κάτι τέτοιο θα υπάρξει. Δύσκολο είναι να πούμε πότε, ωστόσο μπορούμε να μιλήσουμε να απευθυνθούμε σε εναλλακτικού εκπροσώπους της ρωσικής ελίτ στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στο ρωσικό ε, κράτος έτσι ώστε να μην εμπλακούν όλοι στην Ρωσία σε αυτή την υπερεθνικιστική ε, ε, σε αυτό το υπερεθνικιστικό αν θέλετε δίχτυ. ο Πούτιν δημιούργησε την κρίση ασφαλείας και ως Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι μπορούμε να ε, μετριάσουμε, να ελέγξουμε αυτή την κρίση ασφαλείας και να συνεργαστούμε στενά και με άλλους συμμάχους. Με την Ατλαντική Συμμαχία, με τις Ηνωμένε Πολιτείες, τον Καναδά και όλες τις άλλες δυτικές χώρες που έχουν υιοθετήσει την ίδια θέση μέχρι σήμερα όσον αφορά στις κυρώσεις. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι μια μεγάλη μάχη που υψώνεται μπροστά μας είναι η μάχη ενάντια στη ρωσική προπαγάνδα, στην παραπληροφόρηση. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ε, πολεμήσουμε την αμάθεια και την προπαγάνδα που ε, κάνουν. Και σίγουρα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να χαράξουν μια τέτοια ε, πολιτική ε, για να ε, αντιμάχονται τις εσφαλμένες πληροφορίες που διαδίδονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι συγκεκριμένο σήμερα εδώ να λάβω μέρος σε αυτή την ακρόση για την ε, σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία πράγματα. Καταρχήν τις γενικές τάσεις ε, που έχουν κυριαρχήσει στη σχέση αυτή εδώ και πολύ καιρό. Δεύτερον, θα προσπαθήσω να αναφερθώ να πω δύο λόγια για τα θεμελιώδη λάθη που και οι δύο πλευρές, αλλά ιδίω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαπράξει και συνεχίζουν να διαπράττουν όταν ε, εκπονούν και προετοιμάζουν τις, ε, την πολιτική προσέγγιση. Και θα προσπαθήσω τρίτον να πω δύο λόγια για το πώς βλέπω το μέσο μέλλον της σχέσης αυτής. Καταρχήν για τις γενικές τάσεις, ε, το ΖΕΝΙΘ των ε, ρωσοευρωπαϊκών σχέσεων ε, ήταν το Μάιο του 2003 όταν στη Σύνοδο Κορφής στην Αγία Πετρούπολη δεσμεύτηκαν τα μέρη να οικοδομήσουν μία σχέση, μία σιωνή ολοκλήρωσης που ήταν γνωστό κοινά ως κοινή χώρη στον τομέα της δικαιοσύνης, της εξωτερικής ασφάλειας, της παιδείας, του πολιτισμού. Παρ' όλα αυτά αυτό το όραμα δεν υλοποιήθηκε. Το αντίθετο, αρνητικές ε, τάσεις υπερίσχυσαν ε, καθώς ε, έγινε προοδευτικά αυταρχική Ρωσία, μεγάλωνε το κενό των αξιών και αυτό δεν μπορούσε δραστή σε πολιτική ελεξάρτηση, οικονομική σύγκληση δεν λάβανε χώρα και ακόμη και η πρόσβαση της Ρωσίας στον ΠΟΕ δεν οδήγησε στην υιοθέτηση των κοινών οικονομικών κανόνων, απλώς οδήγησε σε νέες διανέξεις. Η εταιρική σχέση για την ενέργεια που αναμενόταν να γίνει ακρογωνίας λίθος μίας αμοιβαία υποφελούς οικονομικής σχέσης με το καιρό γινόταν ολοένα και πιο προβληματική και οδηγούσε τα μέρη στο να τροποποιούν τις στρατηγικές τους ε, και να μην ενδυναμώνουν αλλά αποδυναμώνουν την αμοιβαία εξάρτηση. Η κοινή γειτονή Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας ε, έγινε ουσιαστικά ε, κάτι που αμφισβητεί, το μία επικράτη αμφισβητούμενη και ένα παιχνίδι. Τα συνολικά προβλήματα της συνεργασίας ε, στην ασφάλεια ήταν σπαραδικά και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν μια όθεση που να ωφελήσει θετικά τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και να απομακρύνει τις αμοιβέ ανησυχίες. Κάποιες ε, μεμονωμένες συνεργασίες ε, μεταξύ κάποιων κρατών μελών και της Ρωσίας αναπτύσσονταν καλύτερα από κάποια άλλα, αλλά αυτό δεν μπορούσε να είναι αντιστάθμισμα στο γενική τελμάτωση και στις ε, συγκρούσεις που υπήρχαν γενικά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Με δύο λόγια, η σχέση, ακόμη και αν ήταν οικονομικά σημαντική και για τους δύο, ουσιαστικά σιγά σιγά ε, μετακινούνταν σε μια εταιρική σχέση αναγκαιότητας και όχι επιλογή σε στρατηγική συνεργασία σε άλλους τομείς δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη. Όπως σας είπα, το ζενήκτο το πετύχαμε το 2003, τώρα έχουμε φτάσει το 2015. Αυτές οι τάσεις έχουν ισχύσει, είπα και υπερισχύσει, εδώ και 12 χρόνια. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε και πολύ μεγάλο δικαιωμένο να ισχυριζόμαστε ότι δεν είχαμε προειδοποίησεις, ότι δεν πήγαινε προς σωστή κατεύθυνση αυτή η σχέση. Η κρίση για την Ουκρανία, επομένως, δεν ήταν ένα σημείο καμπής, δεν άλλαξε την τάση, αλλά σε συνδυασμό διαδικασιών που ξεκίνησαν εδώ και πολύ καιρό. Ένας Ρώσος αναλυτής, αναλυτής και λέω ότι είναι Ρώσος, Γιώργη Τιμπόφ, παρατήρησε σωστά ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της Ουκρανικής κρίσης ήταν παραθέτω. Τώρα μπορούν όλοι να σταματήσουν να προσποιούνται. Η Ρωσία μπορεί να σταματήσει να προσποιείται ότι είναι τμήμα τη Ευρώπης και η Ευρώπη να σταματήσει να προσποιείται ότι συμφωνεί. Τέλο τη παράθεση. Δηλαδή με άλλα λόγια, ένα θεμελιώδε πρόβλημα στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία ήταν η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραδεκτεί ότι η στρατηγική εταιρική σχέση είχε σχεδιαστεί και είχε ε, συναυθεί για μια άλλη Ρωσία πιο πλουραλιστική και που θα έβλεπε τη σημερινή Ευρώπη ως ένα μοντέλο ε, που δεν ισχύει σήμερα. επομένω, η αποτυχία της συνεργασίας με τη σημερινή Ρωσία το 2000 ήταν συστημική το μότο που αναλαμβανόταν συχνά ότι θα πρέπει να έχει σχέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία ήταν λανθασμένο και ως προς την αφήγησή του αλλά και ως προς τη στρατηγική. Ως στρατηγική θεωρούσε τις δεσμεύσεις ως στόχο και όχι ως μέσο που μπορεί να λειτουργήσουν όταν συμφωνούν τα μέρη να λύσουν μαζί τα εφιστάμενα προβλήματα. Δεν μπορεί να είναι στόχος. Ω λόγο, στο επίπεδο του λόγου, δημιουργούσε μία εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται περισσότερο στο να βελτιώσει τις διμερεί σχέσει από τη Ρωσία, κάτι που συνεχώ αποδείκνυε. Η Ρωσία που συνεχώς αποδείκνυε ότι δεν ε, ε, ήθελε να δει ε, το δράμα στην κατάσταση που υπήρχε η Ρωσία, αλλά γιατί δεν υπάρχει εδώ κανένα πρόβλημα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντούσε όχι, είναι δραματική κατάσταση και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας. Ε, η εταιρική σχέση, η πρωτοβουλία που λήφθηκε κατά την Προεδρία του Δημήτρη Ντεμιέγκεφ ε, ήταν η καλύτερη απόδειξη της ματαιότητας για τους λόγους ε, της σύναψης σχέσεων. Όμως υπήρχε ικανότητα και της Ρωσίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι με τις Δύσεις να υπολογίσουν τη συμπεριφορά των άλλων στην ε, περίπτωση σύγκρουσης ε, και να αξιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Και οι δύο πλευρές φαίνεται ότι είχαν υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό τους όταν ήταν κοντά η Ουκρανική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβε υπόψη τι ανοιχτέ προειδοποιήσει της Ρωσίας ε, σε σχέση με το ότι θα θεωρούσε την σύναψη συμφωνίας ε, με την Ουκρανία ω μη φιλική πράξη. Τώρα, εδώ δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να έχει υπογράψει τη συμφωνία, γιατί η συμφωνία σύνδεση είναι προ το συμφέρον τη όμω οι Βρυξέλλες θα έπρεπε να προετοιμάσουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το πώς θα απαντήσουν στην αντίσταση της Ρωσίας και ίσως να έχουν στείλει στην ε, Μόσχα ε, ως πρόληψη ένα τέτοιο σχέδιο έκτακτου ανάγκης που θα τεθόταν σε εφαρμογή η δυτική αντίληψη της Ρωσίας συχνά βασίζεται στα οικονομικά της προβλήματα. Αυτή η αντίληψη ουσιαστικά είναι σωστή, αλλά δεν εκτιμά ότι ακόμη και αν είναι οικονομικά αδύναμη η Ρωσία και έχει λίγους πόρους, έχει τις δεξιότητες για γεωπολιτικά παιχνίδια και αυτό της δίνει σοβαρό πλεονέκτημα στη σύραξη έχει λιγότερες δεξιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασιστικότητα. Όμως, επίσης, έχουμε και το θέμα των αδυναμιών που διαστρεβλώνουν την πραγματική εικόνα. Ένας άλλος αναλυτής, ο Σεργέη Καραγκάνεφ, χαρακτήρισε τη Δύση ως ένα πλέγμα χωρίς κατεύθυνση που έχει οικονομικές ανασφάλειες και που ε, δεν έχει όραμα, ε, χάνει από μπροστά του τις ε, ηθικές του πουπιθήσεις αντιλήψεις. Αυτή, σε αυτή την πρόταση όλες οι λέξεις έχουν ένα συγκεκριμένο νόημα. Μιλάει για ένα μόρφωμα χωρίς έναν αρμάτιστο μόρφωμα με οικονομικές αδυναμίες και αυτή η δήλωση συνάδει και με το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας του 2013 που μιλά για την, για την παρακμή της δύση. Το 2014 η Μόσχα δεν περίμενε ότι ε, θα υπήρχε τέτοια μεγάλη υποστήριξη στην Ουκρανία. Όμως οι λόγοι αυτής της λανθασμένης αντίληψης και αυτό υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει. Τα μέσα, στα μέσα του 2000 η Μόσχα έπεισε την Ευρώπη ε, να επιλέξει τα πραγματικά συμφέροντα εναντί των φιλελεύθερων ξένων Το 2008 τα μέλη του ΝΑΤΟ μπλόκαραν την αίτηση της Ουκρανίας και της Γεωργίας για να μην προκαλέσουν τη Ρωσία. Μετά τη ρωσιοργιανή σύραξη η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκατέστησε τις σχέσεις ε, όπως ήταν με τη Ρωσία παρά του ότι δεν είχαν να γίνει σεβαστές οι συμφωνίες πλήρως. Η αντίδραση στην προσάρτηση της Κρυμαίας ήταν ουσιαστικά ρητορική και κάποιες οικονομικές κυρώσεις ε, τέθηκαν με δισταγμούς, ενώ ε, αντίθετα, ακόμη και αν δεν πληρούνταν ε, οι προϋποθέσεις, υπήρχε πολύ μεγάλη πυγμή από την πλευρά της Ρωσίας και τώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Σε αυτές τις συγκυρίες, και φτάνω προς το τέλος, το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον της σχέσης ε, δεν φαίνεται λαμπρό. Η σύρεξη στην Ουκρανία μπορεί να παγώσει, εν μέρη να επιληθεί, αυτό είναι ένα μεγάλο εάν, αλλά αν η ζημιά που έχει γίνει δεν θα ξεπεραστεί γρήγορα. Επομένως, προτείνω το παράδειγμα της στρατηγικής σχέσης ε, θα πρέπει τελικά να αποσυρθεί. Οι σχέσεις ε, συναλλαγίες στην οικονομία πιθανότατα θα διατηρηθούν, όμως σε χαμηλότερο επίπεδο πιθανότατα, συμπεριλαμβανομένων και με μικρότερο βαθμό φιλοδοξιών στο μελλοντικό σχεδιασμό. Και υπάρχουν τρεις λόγοι Καταρχήν, ε, οι τάσει πρώτη σύραξη που ανέφερα στην αρχή θα διατηρηθούν. το χάρη, η διαφοροποίηση της ενεργειακής συνεργασίας συνεχίζεται. Δεν ε, μπορούμε να φέρουμε την κατάσταση πίσω έτσι όπως ήταν πριν 15 χρόνια. Επίσης, σε ένα πιο γενικό οικονομικό επίπεδο, αν η Ρωσία δεν ήθελε να απελευθερώσει τις αγορές της, ε, ακόμη και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΠΟΕ, δεν είναι πολύ πιθανό ότι θα δεσμευτεί πραγματικά σε ένα σύστημα συνολικού ελευθερού εμπορίου από τον Ατλαντικό ως τον Ειρηνικό και θα συμπεριλάμβανε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωστατική Οικονομική Ένωση, ένα θέμα που εξακολουθεί να συζητείται παρά την κρίση. Ο δεύτερος λόγος είναι πιο προφανής η σημερινή οικονομική κατάσταση, η οικονομική κρίση της Ρωσίας την κάνει λιγότερο λογιστική για τις ξένες επενδύσεις. Όσο οι προοπτικές μιας ακόμα ύφεση της πολιτικές σχέσεις και ενώ ακόμη κυκλοκυρώσεων θα παραμείνουν, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικές. Όλα αυτά φυσικά θα αποδυναμώσουν το μηχανισμό ε, των φιλορωσικών λόμπι στις Βρυξέλλες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δεν θα υπάρχουν τόσο διαθέσιμα χρήματα. Γι' αυτό, τρίτον, και αυτό είναι το κύριο, η εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτικών ηγετών, μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύντομα. Αλλά να συμπεράνω λέγοντας και πάλι ότι ακόμη και αν αυτό το σενάριο της ρεαλιστικής οικονομικής επίδρασης που είναι το πιο θετικό σενάριο που μπορώ να προβλέψω αυτή τη στιγμή ε, ζωτικά εξαρτάται από την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος και όχι από το πάγωμα, από το πάγωμά της. Και θα κλείσω εδώ. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φόρμπριχ. Uh, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τιπρόεδρε, Πρόεδρε. Έρχομαι για πρώτη φορά εδώ και είναι μεγάλη μου τιμή. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα πριν από ένα χρόνο. Είπαμε όλοι ότι δεν ήταν ιδεώδης η σχέση μας με την Ρωσία, αλλά κάποιο είδους εταιρική σχέση χρειάζεται. Ε, μπορεί τώρα να είναι κρίση η ουκρανική κατάσταση, αλλά δεν είναι ρήξη. Ερχόμαστε τώρα ένα χρόνο ε, αργότερα, είδαμε τα γεγονότα στην Ουκρανία μέχρι σήμερα ε, και είναι μια ευρύτερη αυτή σύγκρουση με τη Ρωσία. Αντί για εταίρος θεωρείται όλο και περισσότερο πρόκληση η Ρωσία, ε, πρόβλημα ή ε, ακόμα και κρίση. Όταν το καταλάβαμε αυτό, αναρωτηθήκαμε πολύ ποια είναι η ρίζα του κακού. Ορισμένοι θεωρούν ότι το βασικό είναι η προσωπικότητα και η παραφροσύνη του Πούτιν. Ε, άλλοι θεώρησαν ε, ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και ευαισθησία προς τα ρωσικά συμφέροντα και την Ουκρανική πολιτική. Κατά την άποψή μου το κλειδί για να καταλάβουμε το τεράστιο πρόβλημα της Ρωσίας που έχουμε όλοι σήμερα είναι κάπου αλλού. Τι λέω βασικά, ότι έχει μετατοπιστεί η μηχανική στην ε, ρωσική εξουσία 7 χρόνια πριν την Ουκρανική κρίση. Ε, η εξωτερική πολιτική μετά τη μετατόπιση αυτή ε, έχει ως κίνητρα την εσωτερική κατανάλωση, την εσωτερική αστάθεια και κάνουν αυτούς τους λεονταρισμούς προς το εξωτερικό για να κατευνάσουν και να καλύψουν μάλλον την αδυναμία τους στο εσωτερικό. Να το εξηγήσω. Πρώτον, αυτή η μετατόπιση ε, ήρθε με την έλευση του Πούτιν. Όταν ανέλαβε το 2000 για πρώτη φορά αυτό που τον ενδιέφερε κυρίως ήταν να εδραιώσει την εσωτερική σταθερότητα μετά από μια δεκαετία πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ταραχής. Ε, ε, είναι πολύ ε, αυταρχικός, αλλά το, τελικά το επέτυχε με πυγμή. Για να διατηρηθεί η σταθερότητα ε, τον βοήθησε η αύξηση του τιμών του πετρελαίου. Το 2000 ήταν στα 30 δολάρια και έφτασε στα 130 το 2008. Ε, αυτό είναι πολύ μεγάλο εισόδημα και μπόρεσε να το διανύμει και στην ελίτ και σε πολύ πληθυσμό ε, για να ενισχύσει πολιτικά τον τρόπο με τον οποίο ε, διοικούσε, δηλαδή πολιτικά αυταρχικός και οικονομικά ευημερία στη χώρα. Ε, όταν επέστρεψε στην Προεδρία ε, το 12 αυτό απεδείχθη ανεπαρκές. είχε τρωθεί η νομιμοποίησή του και ορισμένοι Ρώσοι είχαν αφυπνιστεί και ήθελαν να αλλάξει η χώρα τους. Δεύτερον, προβλεπόταν ότι ε, τα εισοδήματα δεν θα ήταν σε τέτοια αυθονία όπως το παρελθόν. Η οικονομική ανάπτυξή τους ε, είχε αρχίσει να επιβραδύνεται και ε, οι τιμές του πετρελαίου να πέφτουν όπως και σήμερα φαίνεται. Άρα χρειαζόταν ένα νέο deal και ο Πούτιν ε, το πέρασε από το υλικό στο άϊλο, δηλαδή στο ιδεολογικό. Μίλησε για το μεγαλείο της Ρωσίας, για την αδικία που υπέστη ιστορικά η Ρωσία, τόνισε την ε, υπεροχή τους απέναντι σε μια ε, παρακμάζουσα και ευθύνουσα Ευρώπη και ακόμα και ότι έχει ξεχωριστό πολιτισμό με είδος μεσιανικό και με αποστολή για τον κόσμο και θεωρεί ο Πούτιν ότι έχει ιστορική αποστολή, άρα απαιτεί θυσίε από όλου και όσοι θέλουν, ε, δεν θέλουν να συμμετέχουν θεωρούνται προδότες. Αυτή η σημαντική μετατόπιση έχει πολλές συνέπειε. συνέπειες. Ε, ο Πούτιν για να ε, βασιλεύει και να διοικεί εκεί θα πρέπει μονίμως να υπάρχει κάποια αστάθεια και κάποια σύγκρουση στο εξωτερικό. και η ε, ενίσχυσε τη δημοφιλία του μέχρι 85% και 87% ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις ε, και κατάφερε να επικρατήσει ε, και να κάνει να σοπάσουν και οι επικριτές της επιστροφής του στην Προεδρία. Η ρωσική ελίτ και οι πολίτες έχουν κόστος και από τη ε, διατήρηση νέων εδαφών όπως είναι η Κρυμαία και από τις κυρώσεις. Και πριν ε, ε, επικρατήσει αυτή η ανησυχία και η αμφιβολία χρειάζεται νέα σύγκρουση για αποπροσανατολισμό. Εξού και η Ανατολική Ουκρανία. Και πιο λογικά αυτή η δυναμική χρειάζεται και νέες επελάσεις, Ουκρανία, ενδεχομένως Μολδαβία και Γεωργία, ίσως και Λευκορωσία, ίσως και Καζαστάν, ακόμα και στις βαλτικές χώρες, γιατί όχι. Δεύτερη συνέπεια. Ε, ε, Ρωσία όλο και περισσότερο μοιάζει με μια κοινωνία σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο πόλεμος στην Αλδοδαπή ε, μετασχηματίζει πολλές πτυχές της οικονομίας και της κοινωνίας. Ε, αυτός ο αυταρχισμός και ο έλεγχος πιέζει οποιοδήποτε αντικαθεστωτικό. Καντιφρονούντα που χαρακτηρίζεται πέμπτη φάλαγγα και διοικητικέ πιέσεις υφίστανται τη δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμα και ο τύπος ελέγχεται με την ε, πλήρη κρατική προπαγάνδα. Ε, οι κυρώσεις έχουν απομονώσει τις ρωσικές εταιρείες από τις αγορές και ε, μόνο το ρωσικό κράτος μπορεί να δανείζει τις μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνοντας την εξάρτησή τους από τον Πούτιν και πιέζοντας όσους ήταν πιο ανεξάρτητοι. Και πιο σημαντικό, ο τομέας της ασφάλειας και του στρατού και των όπλων δυνάμεων θα γίνει κρίσιμος. Περικοπές έγιναν παντού, από τις δημόσιες επενδύσεις, τις κοινωνικές παροχές, αλλά όχι στο στρατό και στην αστυνομία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας της χώρας, για το 2015 θα έχουν 10% περικοπές παντού οριζόντιες, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις. Ε, ε, με δύο λόγια, ε, η Ρωσία ε, έχει αλλάξει λοιπόν τώρα το πολίτευμα και το χαρακτήρα της ε, καλλιεργώντας μόνιμες σειράξεις στο εξωτερικό. Ακόμα και με αυτό το μετασχηματισμό της Ρωσίας η απάντηση της Ευρώπης θα πρέπει να είναι πιο μακροπρόθεσμα. Πρώτον, να μεγιστοποιήσει τις ίδιες τις άμυνες της και να ελαχιστοποιήσει τις ευάλωτες πτυχές που προσφέρονται για ανάμειξη της Ρωσίας. Πώς θα γίνει αυτό. Πρώτον, όταν μιλώ για άμυνες δεν εννοώ μόνο στρατιωτικά. Ε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα η Ουκρανία είναι το μέτωπο ε, για την μάχη στην Ευρώπη. Ε, αν επιτραπεί στην Ουκρανία να υποκύψει και άλλες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και ενδεχομένως τα πιο ανατολικά κράτη της Ένωσης θα είναι τα επόμενα. Στην περίπτωση της Ουκρανίας βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε με πολύ διαφορετικό τρόπο και κλίμακα πώς θα βοηθήσουμε. Οικονομικά είναι πολύ μικρή και πενιχρή, πολιτικά ε, δεν της δίνεται δυνατότητα να μπει στην Ένωση και στρατιωτικά απορρίπτουμε ε, την ε, ανάμειξη. Όλα αυτά ε, θα πρέπει να τα ξανασκεφτούμε. Μολδαβία, Γεωργία, ισχύουν τα ίδια, που είναι θέμα χρόνου να μπουν οι Ρώσοι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε επιτυχείς αμυντικές γραμμές με ισχύ σε πολλούς τρόπους. Επίσης, οι βαλτικές χώρες όπου η Ρωσία απειλεί ανοιχτά και επεμβαίνει και το δεύτερο τα Βαλκάνια που είναι ε, πολύ ευάλωτα και στην πολιτική και στην οικονομική επιρροή ε, του Πούτιν όπως έδειξε άλλωστε και η πρόσφατη επίσκεψη του Πούτιν στη Βουδαπέστη θα πρέπει να ενισχύσουμε και ε, ε, την κατάσταση εκεί και να επενδύσουμε. Ε, η βασική μας άμυνα όμως είναι η ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες της Δύσης. Αυτή η ενότητα εμφάνισε αξιοσημείωτη αντοχή το τελευταίο χρόνο που είναι αξιο... αθαύμαστο και αξιέπαινο αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί. Τέλος, πώς θα αποφύγουμε και θα λαχιστοποιήσουμε την ανάμειξη της Ρωσίας με τους γείτονες. Το τελευταίο χρόνο η πρώτη απάντηση ήταν οι κυρώσει, κυρίω οικονομικέ, μετά από μεγάλε αμφιταλατεύσει και δισταγμού. Ε, επέδωσαν, αλλά αυτό σημαίνει και ε, ε, μεγάλη μείωση των τιμών πετρελαίου. Οι κυρώσεις όμως δεν μετέτρεψαν σημαντικά τη ρωσική πολιτική, ούτε πρόκειται γιατί δεν εντάσσονται στη λογική που σας ανέλησα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειωθούν ή να αρθούν οι κυρώσεις, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα νέο σκεπτικό πίσω από τις κυρώσεις. Πρώτον, θα πρέπει να τραγγίζει τη χρηματοδότηση της επέμβασης. Ε, τι σημαίνει αυτό. Η κύρια πηγή τους στα 40% είναι από τις εξαγωγές πετρελαίου. Ειδικά όταν πέφτει το πετρέλαιο θα πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως ή εν μέρη ε, η πηγή αυτή του εμπορεύματος. Επίσης, οι ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, οι ροές κεφαλαίων και μέσω του SWIFT θα πρέπει να ελεγχθούν, οι εισαγωγές και εξαγωγές κεφαλαίων. Ε, για να ε, υπάρξουν πραγματικά εμπόδια και φραγμοί στο ρωσικό τυχοδιοκτισμό οικονομικά. Έχουμε μάθει πολλά τον τελευταίο χρόνο για τους διάφορους τρόπους με τον οποίο επηρεάζουν ε, τις χώρες οι ρωσικές πολιτικές, οικονομικά ή ακόμα και στις επιχειρήσεις ή ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης. Ε, ενώ υπάρχουν μηχανισμοί και αρχές ελεκτικές, δεν έχουν κάνει ε, παρκώς το ρόλο τους. Θα πρέπει και οι αρχές αυτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταλάβουν, ε, να, να τους επισημανθεί ότι ακολουθούν τη ρωσική τακτική. Υπάρχουν και άλλα μέτρα και κυρώσεις που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Η απεξάρτηση από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας και ε, αντιμετώπιση του ρωσικού πληθυσμού, ρωσόφωνου, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τελειώνοντας, μπορεί να φαίνονται αυτά σε ορισμένους τραγικά, δραματικά, σε άλλους ότι ε, είναι κινδυνολογία ή ότι προσπαθώ να θορυβήσω. Αλλά πέρυσι αυτά που έγιναν ε, δεν με κάνουν είμαι Και όλοι ξανά και ξανά έχουμε πάρα πολύ αρνητικά ε, ευνηδιαστεί και ξαφνιαστεί από τη Ρωσία. Και μακάρι να διαψευστώ γιατί και αυτό θα με ανακουφίσει. Ευχαριστώ. Mr. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε εσάς και τον κύριο Λαντσπέρκης για τη διοργάνωση αυτής της ε, πολύ ευπρόσδεκτης συζήτησης για την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία της Ρωσίας. Λίγα σχόλια θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς, συμφωνώ γενικά με το ύφος των ομιλητών οι οποίοι πολύ συχνά αναφέρθηκαν στην έκπληξή μας, υποτίθεται. Εγώ παίρνω τις αποτα... αποστάσεις μου. Εγώ δεν εξεπλάγει και δεν πιστεύω ότι πολλοί στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εξεπλάγησαν με τις εξελίξεις. Καλό είναι να ανακαλύπτουμε τις ψευδεστήσεις του παρελθόντος που είχαμε, ακόμα και αν είναι αργά ή και πολύ αργά. Οι παρουσιάσεις συνάδουν με την πρόσφατη εκπληκτική και πολύ εμπεριστατωμένη έκθεση της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο ε, «Εσφαλμένη ανάγνωση της Ρωσίας στην Ευρώπη». Νομίζω ότι τα σχόλιά τους πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα ερωτηματικό όμως θα ήθελα να βάλω. Πράγματι εξάγουμε συμπεράσματα από την ανακάλυψη των ψευδεστήσεων, των λαθών και των ε, εσφαλμένων αναγνώσεών μας. Εγώ πιστεύω πως όχι. δίστασα ε, κατά πόσο θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Λάντσπεργκης, που είπε ότι δεν μεταμορφώνουμε εμείς τη Ρωσία. Έχει μια θαυμαστή ε, δύναμη να κάνει προβολές σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και με αυτόν τον τρόπο η διεφθαρμένη Ρωσία μας μεταμορφώνει, ελέγχθη. Και αυτό είναι πολύ φρικτό γιατί υπονομεύει την θεμελιώδη παραδοχή ημών ως βασιζόμενων στις συνθήκες. Στις συνθήκες. Θέτει να αμφιβόλω την αξιακή βάση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μέντρας είπε ότι δεν περιμέναμε τα της Κρυμαίας. Κοιτάξτε, εδώ είναι δυτικοευρωπαϊκό το πάνελ σας. Κανείς από εσά δεν είναι από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και μην μιλάτε εξ ονόματος του συνόλου της ΕΕ, γιατί εμείς από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δεν είχαμε ποτέ αυτές τις ψευδεστήσεις. Έχοντας συγκαλέσει την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής, ε, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, εγώ όπου προείδρευα, είχαμε πει τότε ότι ε, σε δύο χρόνια η Κρυμαία θα είναι η επόμενη, γιατί τότε υπήρχε η έφοδος στη Γεωργία. Και εσείς δεν το πιστέψατε. Το 2009 είχαμε επιστολή, τη γνωστή επιστολή διανοούμενων και πολιτικών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ο Χάβελ και ο Βαλέσα την έχουν υπογράψει μεταξύ άλλων, όπου λένε Προσέξτε ότι η Ρωσία είναι απειλή. Ε, γελιοποιήθηκε η επιστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν δόθηκε σημασία στην επιστολή αυτή στην Ευρώπη. Και ε, τώρα παρόλο που είναι αργά αποδεικνύεται αληθινή. Εμείς λοιπόν δεν εξεπλάγημεν, εσείς εξεπλάγημεν από, ε, εκπλαγήκατε από τη Δυτική Ευρώπη. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γιατί χρειάστηκε τόσο καιρό για να καταλάβει κανείς τη Ρωσία, ποιο θα είναι το τίμημα της καθυστερημένης ανάγνωσης και τελειώνω πρόεδρε, ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάναν την εσφαλμένη ανάγνωση τα τελευταία 12 χρόνια πώς θα κληθούν να είναι υπεύθυνοι και δεν θα πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό. Και θα συνεχίσουν με την ίδια γραμμή. Ο χρόνος τρέχει και η Ουκρανία χάνει όλο και περισσότερο έδαφος. Τι διγενέστε να λυθεί αυτό το θέμα, όπως είπε και η κυρία Μέντρας, και να έχουμε αυτές τις δεξιότητες και, και το είπε και ο κύριος Μόσες. Όλα αυτά είναι ε, εξαιρετικά σημαντικά για την ύπαρξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθ' Από τα τρία θεσμικά όργανα εμείς ως πρέπει να είμαστε οι πιο νυφάλιοι, να κάνουμε σωστή διάγνωση των πολιτικών και να μην ε, κρυβόμαστε πίσω από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. I want to be sober in this question, I do not know. Θέλουμε να είμαστε νυφάλιοι σε αυτό το θέμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πρέπει να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών όμως, αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Δύο λεπτά έκαστος για να προλάβουμε. Η κυρία Γκίλ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Βέβαια, άρχισαμε να συγκρίνουμε απόψεις για το ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση απέναντι στη Ρουσία στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης ε, και θα ήθελα να αναφερθώ ε, και στην Βουλή των Ορδών και στην Επιτροπή στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή που είπε ότι ο υπνοβάτης πήγε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανική κρίση και λέει ότι υπάρχει έλλειψη αναλυτικής ικανότητας που αποδυνάμωσε την ικανότητα των κρατών μελών ε, να αναγνώσουν την πολιτική αλλαγή στη Ρωσία για να ε, δώσουν μια αυταρχική απάντηση. Τώρα από τα περισσότερα κράτη-μέλη βλέπουμε πώς μπορεί να υπάρχει σύγκληση και εγώ νομίζω Νομίζω ότι το κλειδί στο να έχουμε μια πιο ισχυρή θέση είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στο θέμα των μυστικών στρατηγικών πληροφοριών. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ανησυχία μου είναι ότι ε, η διαπραγμάτευση της Νορμανδίας ε, την περασμένη εβδομάδα, ήδη καταραίει λέγοντας ε, ότι δεν μπορεί να γίνει απόσυρση βαρέων όπλων καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις. Εσείς τι πιστεύετε για την αποτελεσματικότητα του σχηματισμού της Νορμανδίας και του μηνύματος που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με στην εργασία μόνο δύο κρατών μελών που έχουν επιταχύνει και λυπάμαι πολύ που δεν συμμετέχει το Ενωμένο Βασίλειο ε, καθώς ε, την Κυριακή ε, είπε ότι μπορεί τα ρωσικά αεροσκάφη να χτυπήσουν κάποια επιβατικά αεροπλάνα και είχαμε και άλλα θέματα με τον Υπουργό Άμυνα ε, να λέει ότι η Ρωσία είναι τόσο μεγάλη απειλή για την Ευρώπη όπως το Ισλαμικό κράτος. Ε, πώς ε, λοιπόν εμείς πρέπει να δούμε αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις παραβιάσεις του νερού χώρου και πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις μας είναι σε ένα χαμηλό επίπεδο, σε πολύ χαμηλό, χαμηλό επίπεδο μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και βέβαια είχαμε και τη δολοφονία του Λετιανιένκο από πράκτορες της Καγκεμπέ στη δοκιμά Εθνική Επικράτεια. Αλλά ίσως να έχει δίκιο ο συνάδελφος, ο κύριος Σαρούς Βόλσκι. Ίσως θα πρέπει να δούμε πιο σοβαρά τις απειλές της Ρωσίας και ο Πούτιν ε, ήταν ε, εντελώς ειλικρινής ε, σε αυτά που έλεγε ε, και εγώ νομίζω ότι θέματα που τον ξεφτέλησαν ε, όπως το κοσυφοπαίδιο στο παρελθόν τον ανάγκασαν τα τελευταία χρόνια να σχεδιάζει την εκδίκησή του ε, για να υπάρχει μια αυταρχική καπιταλιστική μεγάλη Ρωσία που θα αντικαταστήσει την πρώην Σοβιετική Ένωση και από ό,τι φαίνεται αυτό τώρα αποτελεί μέρος του νέου σχεδίου η Νέα Ρωσία, το Νοβορόσια. Και ε, επίση αυτό είναι μέρο ε, του ονείρου του Πούτιν ε, και αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθεί και στρατιωτική ισχύ. Η Ρωσία φυσικά δεν έχει σεβαστεί πολλέ από τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει στο διεθνέ δίκαιο, όπω με την προσάρτηση τη Κρεμαία και την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε τι έλεγε κάποτε ε, ο Στάλιν αν ε, θέλουμε να καταλάβουμε τον Πούτιν. Ε, τώρα η διπλωματία είναι για τους δειλούς και ζούμε. Πόσες μεραρχίες έχει ο Πάπας έλεγε ο Στάλιν και Τώρα πρέπει να δούμε πώς ε, θέλουν να δουν ε, να γίνονται τα πράγματα στο μέλλον. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να κλιμακωθούν οι κυρώσεις ε, της Ρωσίας και να χρησιμοποιηθεί και το SWIFT αν παραβιαστεί περαιτέρω η Συμφωνία Μίνσκ 2 και θα έδινα και μέσα στις Ουκρανικές αρχές να υπερασπιστούν τον εαυτό τους αν προχωρήσουν οι αυτονομιστές προς τη Μαριούπολη. η Ελλάδα και η Ουγγαρία δεν θέλουν ε, τις κυρώσεις. Όμως από τη δική μου σκοπιά εγώ νομίζω ότι υπό την ηγεσία του Πούτιν έχει τελειώσει η διπλωματική σχέση. Thank you, Chair. ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν θα σας δώσω τώρα μια συνολική θεώρηση της Ουκρανίας από πλευράς των φιλελευθέρων για να αξιοποιήσουμε την παρουσία των εμπειρογνωμόνων που έχουμε καλέσει για να μας συμβουλεύσουν, να μας βοηθήσουν. Ε, νομίζω ο Πούτιν θα πρέπει να ε, ε, επανέλθει στην νομιμότητα, πράγμα πολύ δύσκολο. Η κυρία Μαντράς είπε, νομίζω, ότι θα πρέπει να κοιτάμε για τη μετά Πούτιν εποχή ε, αυτό μπορεί να έρθει μετά από μία πενταετία και δεκαετία όμως, διότι ο Πούτιν ξέρει πολύ καλά τα παιχνίδια τη εξουσία. Ποια είναι η διαβλή όμως που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα ε, ανεπίσημα, με ποιον, σε ποιον αποτανθούμε στη Ρωσία. Για να δούμε τις κυρώσεις που αυτό συνδέεται με την τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Έχουν τεράστιες επιπτώσεις, αλλά θα ρίξουν τον Πούτιν. Ε, οι εμπειρογνώμονες ε, μας προτείνουν και άλλες κυρώσεις. Υποστήριξη της Ουκρανίας. Εγώ θα ήμουν υπέρ εάν πεθάνει τελείως η συμφωνία του Μίνσκ, καπότι δηλαδή, πράγμα που νομίζω ότι συμβαίνει. Ε, αλλά πώς θα μας συμβουλεύατε, τι να κάνουμε και τι να κάνουμε και για την ε, κοινωνία και τι διδάγματα μπορούμε να βγάλουμε. Ευχαριστώ. I would like to, hear judgment και εγώ θα, ήθελα, να ακούσω την άποψή σας ε, για τη Συμφωνία Μινσκ 2 και θα ήθελα να κατανοήσω πώς βλέπετε ποια είναι η αξιολόγησή σας για τη δυτική προοπτική για τη Ρωσία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Μινσκ 2. Δεν αποτελεί αυτό κατά κάποιο τρόπο τη συνέχιση μιας ανόητης στρατηγικής απέναντι στη Ρωσία. Γιατί εξακολουθεί να βασίζεται στην ιδέα ότι ε, καθόμαστε στο τραπέζι με έναν αξιόπιστο εταίρο, αλλά επιτόπου στην Ανατολική Ουκρανία δεν φαίνεται ότι μπορούμε να βασιστούμε στους ανθρώπους αυτούς με τους οποίους καθόμαστε μαζί και διαπραγματευόμαστε. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πώς θα συνεχίσουμε μετά το Μίνσκ 2, γιατί και εγώ την ε, τελευταία εβδομάδα είδα στην Ανατολική Ουκρανία ότι οι πολίτες αυτό που πραγματικά θέλουν είναι να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, ειρήνη. Και φυσικά οι διεκτικοί πιστεύουν ότι ξέρουν γιατί την απαραίτητη ειρήνη, αλλά οι Ουκρανοί το ξέρουν πολύ καλύτερα γιατί η ειρήνη είναι μια καλή ελεκτική, Αλλά κανείς τώρα δεν καταλαβαίνει τι είναι έτοιμη να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει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 Ένας ομιλητής τόνισε την ανάγκη να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανεξαρτήτους κόστους και αυτό πραγματικά με έκανε να νιώσω φρίκι αν θέλετε γιατί σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τρόπους για να συνομιλήσουμε με την Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως υπογράψαμε συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία και στείλαμε αυτό το χειρό μήνυμα ότι θέλουμε η Ουκρανία να είναι μέλος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή. Ως Κοινοβούλιο δεν έχουμε καν συζητήσει τις ε, ε, επιπτώσεις στο εμπόριο, στη σχετική ε, επιτροπή. Λέγεται ότι η Ένωση δεν έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική και όμως έχει που είναι η επέκταση με κάθε κόστος. Και μάλιστα πρέπει να πούμε για το καθεστώς Πούτιν ότι είτε μας αρέσει είτε όχι ο Πούτιν είναι δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος. Προσωπικά δεν μου αρέσει. Αλλά αυτό είναι μια αλήθεια. Πολύ συχνά λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει την ειρήνη μέσα στην Ευρώπη. Ας μην ευαγγελιζόμαστε όλες αυτές τις νεοφιλελεύθερες φιλοδοξίες. Και νομίζω ότι πολύ εύγλωτα το είπατε εσείς κύριε όταν μιλήσατε για την έκθεση της Βουλής των Λόρδων τονίσατε τη διαφορετική προοπτική που έχουν τα διάφορα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα τραγικό παράδειγμα είναι η κρίση στην Ουκρανία και αυτά δείχνουν γιατί μια κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή ε, πολιτική ασφαλείας δεν μπορεί ποτέ να είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, κύριο Σαφάουζε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, για αυτό ε, το τρίτο σκηνοθετημένο πλήγμα. Και για το αεροπλάνο MH10 περιμένουμε ακόμα τα στοιχεία και τις αποδείξεις. Υπήρχαν δορυφόροι. Είναι στημένο. Το δεύτερο στημένο ήταν η Μαριούπολη όπου σας είχαν πιάσει οι τύψεις πολύ καλά, αλλά ξεχάσατε να μας μιλήσετε για τον Ντονιέσκ ή τον Λουγάνσκ που 10-15 μέρες πριν είχαν βομβαρδιστεί. Και τώρα φέρνετε τρεις προπαγανδιστές που μιλούν με ένα στόμα και μια φωνή, ενώ υπάρχουν επιστήμονες, Έλεν Κάροντοκ, Ζακ Σαπίρ από τη Γαλλία, που σκέφτονται ακριβώ τα αντίθετα και πιστεύουν. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτό το σαμποτάζ της γαλλογερμανικής ειρνευτικής πρωτοβουλίας, σαμποτάζ από Γερμανό αλλά και ε, με την υποστήριξη της Αγγλίας και θέλω να πω ότι η ε, ε, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, οι μεγάλες δυνάμεις δεν σας υποστηρίζουν. Στο όνομα τίνος θα λέτε όλα αυτά, για ποια Ευρώπη, υπέρ ποιας Ευρώπης είστε λοιπόν, την Ευρώπη του μίσου, την Ευρώπη της προδοσίας. Ράδιο Μόσχα λέει ο κύριος Σάρις Βόλσκι. Και ράδιο Ουάσιγκτον κάποιοι άλλοι. Καμιά φορά ο πρόεδρος έχω την εντύπωση ε, ότι όταν δεν ξέρουμε την ουσία υψώνουμε τη φωνή μας. Ιδιαίτερα όταν τα παίρνεις τα λεφτά δανεικά και πρέπει να τα γυρίσεις πίσω. Πλένκοβιτς. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους ομιλητές. Προφανώς ε, υπογραμμίσατε ότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε μάρτυρες για το πόσο μακριά ε, μπορούν να πάνε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία. κύριε Φαμπίκ, ε, είπατε ότι δεν υπάρχουν αυτά που κάνει οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αν ε, τα ποσά που έχουν ε, διατεθεί για την Ουκρανία είναι πολύ μεγαλύτερα ε, συνολικά τα τελευταία 20 χρόνια, αν το εξετάσετε και ακόμη και πολιτικά, απλώ τα μετάμε στο να προσφέρουμε εντάξει, εδώ ισχύει το άρθρο 49 για την Ουκρανία, υπόθηκε αυτό και στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και είπατε ότι στρατιωτικά τι κάνουν τα κράτη-μέλη ότι φαίνεται να είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εσείς ε, τι μας συμβουλεύετε, τι συμβουλεύετε να κάνουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη, αν θεωρείτε ότι αυτά είναι ανεπαρκή για να βοηθήσουν την Ουκρανία να γίνει μια χώρα που θα μπορεί από μόνη της ε, να αποφασίσει για το μέλλον της και την κατεύθυνσή της. Ευχαριστώ.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 Μπορώ να συμφωνήσω με του ε, τρει ομιλητέ και θέλω να του ευχαριστήσω για τη συνεισφορά του Είναι αλήθεια. Όπω είπαν κάποιοι από του συναδέλφου. Ε, σε αυτό τον οίκο υπήρχαν κάποιε φωνέ που έλεγαν ότι η Ρωσία δεν ε, αποτελεί έκπληξη και δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε έτσι. Και πάλι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί εδώ οι οποίοι έχουν εκπλαγεί από τη Ρωσία σήμερα και κάποιοι άλλοι να μιλούν στον Καβαρίτ Μασκβά. Αυτό με φόβησε περισσότερο. Αλλά τώρα, εμείς πρέπει να δούμε το εξής. Έχουμε την ε, ε, προσάρτηση της Κρυμαίας. Είναι το ρωσικό στυλ. Έχουμε μια συμφωνία η οποία προσπαθεί να ευλογήσει ε, την προσάρτηση, την κατοχή και επίσης έχουμε και κάποιες άλλες προκλήσεις που προσπαθούν να εξηγήσουν περαιτέρω την επέκταση Ρωσίας. Έτσι ονομάζεται το παιχνίδι και στην περίπτωση μιας ε, συμπεριφοράς χιτλερικού τύπου εμείς ε, θέλουμε να απαντήσουμε με ένα στυλ Τσάμπερλεν και ξέρουμε ε, την ιστορία όταν Τσάμπερλεν συμπεριφέρθηκε στη Γερμανία ότι έκανε είχαμε το δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο και Πολύ μου αρέσουν ε, όλοι όσοι και θα ήθελα ε, όσοι εκφράζουν κάποιες αφελείς τάσεις εδώ να δουν την ιστορία και να καταλάβουν τη σοβαρότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να έχει περαιτέρω αμυντικές ικανότητες ε, παράλληλα με το ΝΑΤΟ και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να καταπολεμήσει τη ρωσική προπαγάνδα και τη χρηματοδότηση των κομμάτων και των ΜΚΟ που γίνεται τώρα ε, το πέμπτο τάγμα ε, σε ρωσικό, την πέμπτη φάλαγγα σε ρωσικό στυλ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Βανόρδεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι θέμα ΕΕ Ρωσίας, αλλά δυτικών δημοκρατιών και Ρωσίας. Και αν θέλετε, ως πρώην ε, μαχητής του ψυχροπολεμικής της ψυχροπολεμικής εποχής καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα για τη Ρωσία. Η Ρωσία καταλαβαίνει τη δύναμη, θα εκμεταλλευτεί το διέρη, τα διαιρέσεις και καταλαβαίνει την αξία του εκφοβισμού της δυτικής κοινή γνώμης και θα μάθει από τα βήματα που θα κάνουμε στην πράξη κατά πόσο είμαστε σοβαροί και έχουμε πραγματικές κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν θα περάσουμε. Και όλα αυτά υποκρύπτουν τη στρατιωτική και οικονομική της αδυναμία. Ερωτώ τους ομιλητές, πιστεύετε ότι ο Πούτιν έχει σαφές στρατηγικό πρόγραμμα και αν ναι, ποιοι είναι οι πραγματικοί του στόχοι ή το μόνο που κάνει είναι να αρπάζει τις ευκαιρίες που, ε, όσο αυτές εμφανίζονται μπροστά του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Αουστρεβίσιους στρατιωτικά επιθετική, οικονομικώς αδύναμη και πολιτικά αυταρχική. Αυτή είναι η Ρωσία που αντιμετωπίζουμε ως φαινόμενο τώρα. Και όταν ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη η Ρωσία, δεν συζητούσαμε μεταξύ ημών και ημών, με ήττα και ύψιλον αντιστοίχω, αλλά μέσα στι κοινωνίε μα συζητούσαμε. Μέρο του κοινοβουλίου αυτού δείχνει την πλήση εγκεφάλου την οποία κατάφεραν να κάνουν οι Ρώσοι τι τελευταίε δεκαετίε. Η σημερινή Ρωσία, η φετινή Ρωσία, το Μάιο, άρχισε να μιλάει γαλλικά, τον Ιανουάριο άρχισε να μιλάει γερμανικά και ήδη μιλάει αγγλικά και ισπανικά έτσι έχει το πάνω χέρι για να αποκτήσει πρόσβαση στη δική μας κοινή γνώμη, να του κάνει πλήση εγκεφάλου των τους ευρωπαϊκούς λαούς και να παραπληροφορήσει. Ερωτώ λοιπόν τα μέλη του πάνελ, ποια είναι η άποψή τους. Τι και πώς θα πρέπει να το κάνουμε, τι θα πρέπει να γίνει για να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας από αυτό τον πόλεμο πληροφοριών, γιατί η Ρωσία για πάρα πολλά χρόνια είναι εναντίον μας. Ευχαριστώ. <clears throat> Κύριο Πάσκο, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ενότητα στην ανάλυση των τριών συναδέλφων που ήρθε εδώ είναι κάτι που το βλέπω ως εξή. Επικεντρώνεται γύρω από το γεγονός ότι το καθεστώς στη Μόσχα είναι ο πραγματικός επέτειος και αυτούργός των όσων συμβαίνουν και θα πρέπει στρατηγικά να το αντιμετωπίσουμε. Και το ερώτημα είναι, είναι δικτάτορο ο κύριος Πούτιν ή Ιωνί δικτάτορ ή έτσι θα γίνει ε, ή μπορεί να ανακληθεί στην τάξη, μπορούμε αυτό να το αποτρέψουμε. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά το θέμα είναι πώς θα διηθηθεί αυτή η κοινή θέση του ακαδημαϊκού κόσμου, του πανεπιστημιακού, για να φτάσει στο επίπεδο της λήψης των αποφάσεων. Θα πω δύο λόγια μόνο και θα κλείσω. Πρώτον, ένας από τους λόγους γιατί που μπήκαμε εμείς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να απαγκιστρωθούμε από αυτή τη ε, φαιά περιοχή, γκρίζα ζώνη, ανάμεσα στις ανατολικές και δυτικές δυνάμεις. Πάντα ε, ε, ήταν εις βάρος μας αυτή η διελκυνστίδα. Και τώρα που ανήκουμε σε αυτούς τους θεσμούς, σε αυτούς τους οργανισμούς, ελπίζουμε να έχουμε ξεφορτωθεί αυτό το μοτίβο 100-150 ετών ευρωπαϊκής πολιτικής που αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην Ουκρανία. Δεύτερον, οποιαδήποτε προσέγγιση έχει κάποιος για τη Ρωσία, ραπροσμόν κτλ. Ε, εγώ νομίζω ότι έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στη Ρωσία και στις ιδέες που την εμφορούν και θα πρέπει στρατηγικά να εξασφαλίσουμε παράλληλα με οποιαδήποτε προσέγγιση ή ουδήποτε στο μυαλό του για τη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά και τελείωσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόκληση που θέτει ο Πούτιν στην Ευρώπη. Είναι μικροπρόθεσμο, γι' αυτό και εμεί πρέπει να δώσουμε μικροπρόθεσμη απάντηση. Δεν μιλάμε μόνο για τα διάφορα συμβάντα στην Ευρώπη. Έχουμε κάποιες χώρες που θέλουν να κάνουν τη δυτική επιλογή, αλλά πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει στο ευρωσιατική επικράτεια ε, που ε, ε, οικοδομούν και κάποιε στρατηγικέ κάποιες στρατιωτικές δομές. Ε, τέτοιες χώρες όπως ε, η Αρμενία ε, βρίσκονται σε μια εμπλοκή για την δυνατότητα να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, το όπλο των κυρώσεων και πρέπει να σκεφτούμε ποια απάντηση θα δώσουμε. Καταρχήν πρέπει να ενδυναμώσουμε την άμυνά μας. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τη Ρωσία να συνειδητοποιήσει ποια θα είναι η απάντησή μας αν ληφθούν πιο επιθετικά βήματα. Επίσης πρέπει να έχουμε και την δυνατότητα να ενταχθούμε ενταχθεί ταχαίως η Γεωργία στο ΝΑΤΟ και να ενδυναμώσουμε την ε, άμυνα των ε, βαλτικών χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία επίσης. Ε, θα πρέπει να έχουμε συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διπλωματική απάντηση όπως παραδείγματος χάρη στο ουκρανικό ζήτημα να υπάρξει αποστολή ρηνευτικών δυνάμεων, κάτι που ζητάει η Ουκρανία. Η Ρωσία λέει ψέματα και γι' αυτό είναι λυπηρό που το κοινοβούλιο μας και κάποιοι από την Επιτροπή μας δεν ήθελαν να υποστηρίξουν τη συζήτηση για την 70η επέτειο της εγκατάλειψης των ανατολικών χωρών στη Γιάλτα. Εγώ νομίζω ότι αν τα λύσουμε όλα αυτά δεν θα υπάρχει πλέον παράθεση με τη Ρωσία. Μικρόφωνο, ε, πρέπει να φύγουν σε λίγο οι διερμηνείς και θα πρέπει να μιλήσουμε όλοι αγγλικά. Α, από αυτή τη στιγμή και μετά σχολάνε οι διερμηνείς και θα συνεχιστεί στα αγγλικά η συνεδρίαση the arrangement between you and your translators is something bilateral, it's not multilateral. Α, τα θέματα που έχετε εσείς με τους διαρμενίστες είναι διμερεί, όχι πολυμερεί. Μάικρο. Jaz ne pričakujem aplauza po današnji razpravi in sploh mislim, da so aplauzi predvsej neokusna zadeva, kadar gre za razprave o tako resnih zadevah, kot je vprašanje vojne in miru Mislim, da je zelo dobro bilo zadeto, ko je nekdo rekel, da mi ne znamo predvidevati stvari, da smo vedno znova presenečeni. Presenečeni smo bili mi, Zahod, v Afganistanu, v Iraku, v Libiji, povsod smo presenečeni in na koncu smo bili presenečeni v Libiji, v Ukrajini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 po mili volji okupira teritorij druge države in vojaško intervenira. vendar pa mislim da bi morali kadar se pogovarjamo zlasti o ukrajini nekoliko pobrskati po svojem spominu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 je pa nekoliko drugačen od, od odnosa držav, ki so bile neposredno prizadete z sovjetsko brutalnostjo, okupirane in, in doživljale to, pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. Vem, da mi boste vzeli besedo,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 sedenju za mizo in pogajanju ni. Hvala lepa za pozornost. Jaz sem se prijavil za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Me me too, Mr. So, Mrs. Yakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. I have two questions. First, background